Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, έχω μία δήλωση να ε, διαβάσω. Θα θυμάστε ότι ο πρόεδρος κατά τη συνεδρίαση στις 11 Μαΐου 16 επέβαλε μια κύρωση στο συνάδελφο Συναδεινό γιατί έκανε απαράδεκτες ε, δηλώσεις για τον τουρκικό πληθυσμό κατά την Ολομέλεια της 9 Μαρτίου. Στο Προεδρείο τη Δευτέρα 6 Ιουνίου με την ένσταση του κυρίου Συναδεινού και ομόφωνα αποφασίσαμε να ευεβεβαιώσουμε την απόφαση του Προέδρου. Η κύρωση είναι η αφαίρεση 10 ημερήσεων ε, αποζημιώσεων από τον κύριο Συναδεινό και πληροφορήθηκε γι' αυτό χθες. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Όχι, όχι. Έχει λήξει η διαδικασία. Οι συνάδελφοι, ο συνάδελφος την